είναι κάτι το οποίο μας ε, σοκάρει ως κοινοβούλιο και επιπλέον ακούμε δυσάρεστα νέα και από το Ιράν. Ανησυχούμε για την καταδίκη σε θάνατο των αντιφρονούντων.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 για την υπογραφή των ε, πράξεων που έχουν ε, υιοθετηθεί υπό την κανονική νομοθετική διαδικασία. Θα υπογράψουμε